Θα συνεχίσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. 38 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για επεξηγήσεις ψήφου. Ας περιμένουμε τρία λεπτά για να μπορέσει να κατακαθίσει λιγάκι η κατάσταση στην Ολομέλεια, να μπορέσουν να φύγουν όσοι θέλουν να φύγουν.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 Όσοι φεύγουν παρακαλώ να το κάνουν ώστε να τον πιο γρήγορα και ήρεμα και σιωπηλά γιατί έχουμε πάνω από 40 επεξηγήσεις ψήφου. Ο κάθε συνάδελφος θα έχει ένα λεπτό όπως πάντα. Πρώτα για την έκθεση Μπέγκε κινητοποίηση του εργαλείου ευκαμψίας ο κύριος Σιλβέστρος έχει το λόγο πρώτα. Grazie Presidente. L'attivazione dello strumento Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ε, έγκριση του μέσου ευελιξία ε, δείχνει ότι περισσότερο χρειάζεται ευελιξία ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό, γιατί υπάρχουν ε, πολλές περικοπές σε διάφορες γραμμές του προπολογισμού, ενώ η κατηγορία 1α και η 4 δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς καθορισμένες προτεραιότητες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου Εν τω μεταξύ, το μέσο ευελιξίας χρησιμοποιείται για να δώσει 175 εκατομμύρια ευρώ στην κατηγορία 1α και 267 εκατομμύρια ευρώ στην ε, κατηγορία 4. Η χρήση ε, αυτού του μέσου ευελιξίας για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής 2020 ε, σημαίνει 242 εκατομμύρια επιπλέον και γι' αυτό και ψηφίσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Δανιέλ Χάναν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, διερωτώ με από πού προέρχεται αυτή η ιδέα ότι ο τρόπος για να πλουτίσει κανείς είναι να παίρνει ενισχύσεις, επιδοτήσεις. Δεν αληθεύει ούτε για άτομα ούτε για επιχειρήσεις ούτε για χώρε. Ε, αν ήταν αλήθεια, η Ελλάδα θα ήταν τώρα ζάμπλουτη ε, και οι Έλληνες. Ε, και οι Γερμανοί διαμαρτύρονται, λέει, για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα ενισχύσει στην Ελλάδα. Όμω, όπως το βλέπουμε, αυτό είναι βλαβερό για το ΑΕΠ και αυτό ισχύει γιατί όπως μεταξύ ατόμων έτσι και μεταξύ κρατών ο κόσμος αρχίζει να ρυθμίζει τα θέματα του ε, προσπαθώντας να γίνει επιλέξιμος για να πάρει χρήματα. Το ίδιο γίνεται και με τα κράτη λοιπόν, η ίδια αρχή. Υπερβολική παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αίτιο των προβλημάτων μας και δεν πρόκειται να είναι η λύση. Η την κοινή έκθεση της κυρίας Μπαρζάνη και του συναδέλφου Χωζέ Μανουέλ Φερνάντες έχει τώρα το λόγο ο συνάδελφος Άσλι Φόξ. Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εγκρίνουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2012, μια αύξηση στι πιστώσει πληρωμών κατά 2%. Αυτό είναι μια νίκη για τα κράτη-μέλη και για του καταναλωτέ έναντι του Κοινοβουλίου αυτού και τη Κομισιόν. Όσο δύσκολο να το πιστέψει κανεί, η Κομισιόν ζήτησε μια αύξηση 4,3% και το Κοινοβούλιο ήθελε 5,3%. Όλα αυτά σε μια στιγμή που οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τους φόρους και να μειώσουν τις δαπάνες σε εθνικό επίπεδο. Μήπως υπάρχει καλύτερη ένδειξη του πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, πόσο δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ακόμα και 2% για μένα είναι πάρα πολλά θα πρέπει να περικόψουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσουμε το άχθος των φορολογουμένων. Αντί να ζητά αύξηση κονδυλίων, η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με σοφροσύνη τα χρήματα που παίρνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζορτζ Λάιον. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να υποστηρίξω τον προπολογισμό όπως ενεκρίθη σήμερα. Εγώ συμφωνώ και υποστηρίζω τη Συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2012. Πρέπει να υπάρξει και κάποια αντανάκλαση των, αυστηρών περικοπών που έχουν γίνει στα εθνικά κράτη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέρος στην κοινή προσπάθεια μεγαλύτερη αυστηρότητα και λιτότητα και πιο μεγάλη υπευθυνότητα στι δαπάνε. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την αύξηση του προεπολογισμού μόνο κατά 2% που είναι πολύ λιγότερο από αυτό που είχε ζητήσει καταρχήν η 4,3% και 5,3% από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν σωστή λύση. Αυτό είναι ο μόνο ρεαλιστικό τρόπο για να προχωρήσουμε στα επίπεδα του προπολογισμού. Χαιρετίζω λοιπόν την υποστήριξη τη θέση του Κοινοβουλίου και χαίρομαι το, το γεγονό ότι υπήρξε μια συμφωνία. Ήταν καλή απόφαση και η οποία δίνει καλή εικόνα για το Κοινοβούλιο μας. Ευχαριστώ. Δίνει... Έχει το λόγο ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει το ρόλο του όπως έπρεπε. Μέσα στο σωστό χρονικό διάστημα έχουμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Όλα πήγαν καλά. Αυτές είναι οι καλές ειδήσει. Τα αρνητικά νέα είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη συνέχεια δίνουν νέα καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του ζητούν να τα εγκρίνει, αλλά όταν πρέπει να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα εγχειρήματα δεν συμφωνούν να τα χρηματοδοτήσουν. Δεν δίνουν πρόσθετα κονδύλια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε στο μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι να παίρνει όλα τα καθήκοντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρί να χρηματοδοτούνται και να πρέπει να κόψει το λαιμό του να τα χρηματοδοτήσει. Γι' αυτό εγώ έχω κρατήσει στάση αποχή στην τελική ψηφοφορία, γιατί πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ληφθεί στα σοβαρά. Τονίζω όμω ότι ανέλαβε πλήρω τι ευθύνε του σε σχέση με την ψήφιση. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο και πάλι στον κύριο Σιλβέστρη. Κύριε Πρόεδρε, μετά από 15 ώρες επικοδομητικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώνεται ε, η, διαπραγμα... η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ε, με την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου του περασμένου Ιουλίου. Ωστόσο, Είμαστε πάνω από τι ε, προτάσει του Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όταν ε, καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε περιθώριο λιγμό για τι ιστώσεις ε, υποχρεώσεων, λαμβάνοντα υπόψη πω τα κράτη-μέλη είχαν δυσκολίε και στου εθνικού του προπολογισμού. η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεσμεύτηκε για την ανταγωνιστικότητα και τι εξωτερικέ σχέσει. Γι' αυτό και στηρίζω αυτό το προπολογισμό του 2012 που δεδομένων των δυσκολιών των οικονομικών και των δημοσιονομικών μπόρεσε να να βρει μία λύση ε, για να δώσει πνοή στην ανταγωνιστικότητα, στις καινοτομίες και στις επενδύσεις που είναι χρήσιμες για την ε, ευρωπαϊκή ανάκαμψη. Επίσης, προ... συμφωνία σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας εντός των προθεσμιών που προβλέπονται. Ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστη. Τώρα για την έκθεση του κυρίας Μοντρεμός, ο ε, Γκουτιέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το 2010 ζούμε, ειδικά στην Ευρωζώνη, μία άνευ προηγουμένου κρίση ε, του δημοσίου χρέους στην πιο πρόσφατη ιστορία μας και δείχνει πόσο ασθενή είναι τα μέσα που έχουμε στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία των λεγόμενων αγορών. Ένα από τα μέσα αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πολιτική φιλοδοξία κατά την άποψή μου σαφώς ανεπαρκεί για την καταπολέμηση της κρίσης και την αναζωγόνηση της ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη, μείωση των επιτοκίων έχουν κάνει άλλες κεντρικές τράπεζες για να ενισχύσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Και κατά δεύτερο λόγο, ε, ε, ε, πενέβησαν στη δευτερογενή αγορά μόνο όταν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να προστατεύσουμε το νόμισμά μας με μια τράπεζα τελευταίας καταφυγής, ε, αλλά που να δρά γρήγορα και αποφασιστικά. Και ε, αυτό εξηγεί και ε, τις απαιτήσεις που έχουμε για το μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Μπασέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή, γιατί η σταθερότητα των χρηματαγορών πρέπει να επέλθει κάποια στιγμή. Χρειάζεται η Ευρώπη ένα κατάλληλο πλαίσιο για την οικονομική της πολιτική έτσι ώστε τα δημόσια χρέη να περιοριστούν. Ε, χαιρετίζω την ενεργή ε, δράση ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται οι μέθοδοι αξιολόγησης. Επίσης, να ενημερώνονται καλύτερα οι τράπεζες ε, σχετικά με τα αποθεματικά της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Είμαι υπέρ ε, της μακροοικονομικής εποπτείας για τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης και εκείνων που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Χρειαζόμαστε μια ισόρροπη και επικοδομητική στάση της ΕΚΤ απέναντι σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, διαχειρίζεται τα μέσα που έχει στη διάθεσή της με τρόπο υπεύθυνο. Και μάλιστα μπορεί να τυπώνει και να κόβει χρήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκο. Και πάλι ο κύριος Σιλβέστρης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που μας παρουσίασε σήμερα η κεντρική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει στοιχεία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το 2010 κατέγραψε μείωση το, ε, σε τεράστιο ποσοστό αυτό λόγω της ε, κρίσης. Ε, αυτό και επηρεάζει τόσο το ευρωπαϊκό σύστημα όσο και, το... και επηρεάζεται και από το αμερικανικό σύστημα. Το Διευθυντήριο αποφάσισε να μεταφέρει τις 31 Δεκεμβρίου 2010 1.300 εκατομμύρια, 1 ε, εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ε, έκλεισε λοιπόν το 2010 με ένα περίσευμα το οποίο το Συμβούλιο αποφάσισε να μοιράσει στις κεντρικές τράπεζες της ε, Ευρωζώνης. Αυτό προορίζεται στην παροχή πιστώσεων και εξετάζεται ετησίως. Έτσι έχουμε τον ε, φάκελο, το χαρτοφυλάκιο μάλλον, το οποίο η κάθε μία τράπεζα θα πρέπει να, προσδί, να αποδίδει στην κεντρική τράπεζα και να καθορίζεται έτσι η νομισματική πολιτική μέσα στο πλαίσιο των ομολόγων και στο πρόγραμμα της αγοράς. Κύριε Σιλβέστρης, έχετε χρησιμοποιήσει διπλάσιο χρόνο από το κανονικό χρόνο αγόρευσης. Επομένως, δεν θα σας δώσω το λόγο στο επόμενο θέμα. Στην επόμενη έκθεση, της οποίας την πατρότητα αρνήθηκε ο κύριος Γκέρνς για την χρηματοδότηση των συμπληρωματικών μέτρων για τον τομέα των μπανανών. Έχει το λόγο ο κύριος Χάντς Πέτερ Μάιερ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ψήφισα κατά της ε, τροποποίησης των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα, γιατί για αυτή την ε, έκθεση δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η συνθήκη της Λισαβόνας και η διαδικασία της. Δίνει τη δυνατότητα η τροποποίηση αυτή να μπορεί να παίρνει αποφάσεις μόνο το Συμβούλιο για 10 σημαντικές χώρες ΑΚΕ. Δεν υπάρχει ούτε μια νομική ούτε μια πολιτική αιτιολόγηση γιατί το Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να έχει καμία συμμετοχή στην διαδικασία ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό ιδιαίτερα είναι αντίθετο με το, την ανάγκη το Κοινοβούλιο να, να διατηρεί τις αρμοδιότητές του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να δίνονται κονδύλια στην πολιτική αυτή χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να θέσει σε εφαρμογή τις πράξεις αυτές μόνο μετά το 2013. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι ισότιμες με το Κοινοβουλίο και δεν πρέπει να τις απο, απορρίπτουμε εμεί οι Ο κύριο Κάσμαν έχει τον λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλλον τη, του, της εργατικής ομάδας εμείς υποστηρίξαμε υπέρ αυτής της έκθεσης γιατί δίνει εγγύηση, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα υπάρξουν εναλλακτικέ λύσεις χρηματοδότησης. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τις μάχες μας για τις εξουσίες μας στην πλάτη των φτωχότερων του κόσμου. Εμείς ως ε, τμήμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής τονίσαμε την ανάγκη να είμαστε αξιόπιστοι, αξιόπιστοι εταίροι. Δεν πρέπει λοιπόν να χαθεί αυτή η δήλωση η οποία ενεκρίθη σαν τμήμα του πακέτου και περιλαμβάνει μια σωστή πράξη του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, τις μελλοντικέ πράξεις χρηματοδότησης. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δεχτεί περισσότερο στον τομέα αυτό, αλλά τονίζουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν προκαταλαμβάνει μελλοντικέ συμφωνίε και στο μέλλον θα πρέπει οι κατεξουσιοδότηση πράξη πάντα να περιλαμβάνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριο Σιλβέστρη. Μισό λεπτό. Έχετε μισό λεπτό για να με λάβετε το λόγο. Ναι, 10 δευτερόλεπτα το Ευρωκοινοβούλιο είναι έτοιμο να δεχτεί το συμβαστικό πακέτο εφόσον είναι σύντομη η υπολοιπόμενη διάρκεια των μέσων. Όμω, λόγω του Συμβουλίου δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το κείμενο του μέσου, ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου στι στρατηγικέ επιλογέ, για τι οποίε η ισότητα μεταξύ των ε, διαφόρων νομοθετών είναι πολύ σημαντική. Περνάμε στην έκθεση του κ. Σόλτ για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Κύριο Σιλβέστρης έχει πάλι το λόγο. Προέκυψε μία διαφορά απόψε ανάμεσα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά την έγκριση των πολιετών προγραμμάτων συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων κατέστησε απαραίτητη στη συνδιαλλαγή που οδήγησε στι τέσσερις συμβαστικέ προτάσεις. Στην περίπτωση του μέσου με τις βιομηχανοποιημένε χώρες, η τροποποίηση είχε στόχο να επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο των προγραμμάτων στις χώρες που είναι ακόμα ε, μέσα στο πλαίσιο του, μέσου, του παραδοσιακού μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία. Θέλουμε να συμπεριληφθούν εδώ οι συγκεκριμένες ε, οικονομικές ε, τα κονδύλια μάλλον που προορίζονται για την κάθε χώρα. Για το Συμβούλιο αυτές οι ενδείξεις δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνουν ε, την, ε, τα κονδύλια που θα δοθούν στις συγκεκριμένες χώρες. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστρης και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση της, της κυρίας Γκάλ και Λοχμπίλερ για το χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων παγκοσμίω. Και πρώτα έχει το λόγο ο κύριος Νικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι θεμελιώδεις αρχές τις οποίες εδράζεται και ε, βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ενισχύεται αυτό από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζεται οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα προστατεύει για ε, ε, έναντι τρίτων χωρών. Yeah. Το νέο ε, νομοθετικό πλαίσιο, η χρηματοδότηση ε, του μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι πολύ σημαντικό και με διαφάνεια και καλύτερο τρόπο διαχειριζόμαστε τα κοινοτικά κονδύλια. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δημοκρατική νομιμότητα γιατί εκπροσωπεί λαούς. Γι' αυτό η θέση του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα ζήτημα αρχής. Ευχαριστώ. Gracias. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σιλβέστρης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο που το οποίο ψηφίζαμε αποτελεί ένα μέσο, μάλλον ε, θεσπίζει ένα μέσο για την προπαγή τη δημοκρατία και των δικαιωμάτων ανθρώπων και συμβάλλει έτσι στην ανάπτυξη τη Δημοκρατία και του κράτου δικαίου, το σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να εξασφαλίσουμε την ε, αποδοτικότητα το, αυτού του μέσου θα υπάρξει στενός συντονισμός ανάμεσα στις δραστηριότητες της Κομισιόν και αυτές των κρατών μελών προωθείται περισσότερο σεβασμό στις δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες όπου αυτά απειλούνται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ζητούσε μηδενική ανεκτικότητα απέναντι στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι ανεξισχύω τη συνθήκη Λισαβόνα έχει καταστήσει το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων νομικώ δεσμευτική, μετατρέποντα τι βασικέ αξίε σε συγκεκριμένα δικαιώματα. Αυτή η σημερινή ψηφοφορία προσφέρει ένα παράδειγμα ισχυρό και συγκεκριμένο και μια νομική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστρη. Ο συνάδελφος Χάναν ε, έχει το λόγο. Δύσκολο κύριε Πρόεδρε να μην διασκεδάσει κανείς από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οποίοι καταδικάσουν την απεικιοκρατία και τον υπεριαλισμό χαίρονται να υπογραμμίσουν, να υποστηρίξουν αυτή την ιδεολογία όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα όπως οι τοπικές ε, αντιπροσωπείες, τα θέματα της αντισύλληψης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Από πού νομίζετε ότι βρίσκουμε όλα αυτά τα χρήματα, αν δείτε αυτούς που βρίσκονται στις πιο εύρωστες χώρες, όταν βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι στην κατάρρευση, γιατί να ακολουθήσουν τα δικά μας ε, μηνύματα. Η έκθεση Γκέι Μίτσελ για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο κύριος Σιλβέστρης και πάλι. Ο βασικό γενικό στόχο τη συνεργασία για τι αναπτυξιακέ συνεργασίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δώσει ε, και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και καθώς και την επιδίωξη των στόχων της χιλιετίας καθώς και η προστασία της δημοκρατίας, της, συστής διακυβέρνησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η στήριξη που δίνεται μέσω του μέσου, Μηχανισμού Χρηματοδότησης ενεψυχικής Συνεργασίας προωθεί ε, γεωγραφικά προγράμματα στη βοήθεια στην Νότια Αφρική και στις 47 αναπτυσσόμενες χώρες στη Λατινική Αμερική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ε, η δήλωση δύο της χιλιετίας αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς, στόχος το οποίο είναι η εξάλληψη της απόλυτης στόχης, δηλαδή των ανθρώπων που ζουν με κάτω από ένα δολάριο το ημέρα μέχρι το 2015. Βασική αναφορά για όλες τις χώρες. Ένα τρίτο της, της αναπτυξιακής βοήθειας της Ιταλίας είναι ε, στα χέρια της, της Κομισιόν των Βρυξελών. Γι' αυτό και είμαι υπέρ αυτής της διάταξης, αυτού του μέσου. Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση του κυρίου Σίμψον για τι στατιστικές καταγραφέ των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και έχει το λόγο ο κύριο Σιλβέστρη. για επεξήγηση ψήφου. Εγώ θα μιλήσω εδώ μία φορά, όχι δύο φορές, μία φορά όπω έλεγε στην οθόνη το να ορίσουμε νέες συνθήκες ε, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και στην Κομισιόν. Αυτό είναι το νόημα του άρθρου 290 για τις συνθήκες για τη λειτουργία της, εσωτερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικές αυτές οι ισορροπίες και πρέπει να υπογραμμίζονται. Εξάλλου η άσκηση των κατεξοδότησεων ε, αρμοδιοτήτων δεν σημαίνει ε, ότι δεν ελέγχονται. Ε, τώρα, όσον αφορά τον κανονισμό για τις στατιστικές για τον τουρισμό, η Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών θα πρέπει να ψηφίσει τροπολογίες σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχει αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν μια καλή βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Κομισιόν del... Ευχαριστώ κύριε Σιλβέστης. Περνούμε στη σύσταση του συναδέλφου Σφόμποτα για τη συνθήκη προσχώρησης ε, της ε, ε, κρατικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη έχει το λόγο η κυρία Ελένα Πασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα φυσικά την έκθεση αυτή, διότι η υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ιστορική στιγμή για την Κροατία. Εγώ επιθυμώ σταθερότητα στα Βαλκάνια. Η προοπτική ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης γίνεται πραγματικότητα και ε, οι κόποι ε, τους πιάνουν τόπο. Αυτό όμως δεν είναι το τέλος μιας προσπάθειας. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειές μας στη δικαιοσύνη για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν και τα ναυπηγεία, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον χρειάζεται με τρόπο αντικειμενικό ε, καταγραφή των προόδων της Κροατίας. Ε, πολλό δε μάλλον που για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία διατηρήθηκε ο μηχανισμός επιτήρησης και ε, παλήθευσης. Επίσης θα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη έτσι ώστε η διαδικασία κύρωσης να στεφθεί με επιτυχία. Η ένταξη της Κροατίας αποτελεί καλή ευκαιρία για να αρχίσει και πάλι μια εκστρατεία επικοινωνία σε όλα τα κράτη-μέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Ο κύριος Σιλβέστρης. δήλωση της ανεξαρτησίας και 8 ε, χρόνια μετά από την πρώτη αίτηση της ε, Κροατίας για να εισχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρώσει μια ιστορική διαδικασία η Κροατία και το είδαμε με πόσο ενθουσιασμό ε, χειροκρότησαν οι ευρωβουλευτές του εκπροσώπους του Κροατικού Κοινοβουλίου ε, έτσι ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις ε, έξι ετών και προετοιμασίες πολλών ετών που προώθησαν ε, τη πολιτική και πολιτιστική αλλαγή στις χώρες, στην χώρα αυτή. Εμείς θα ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα σε σχέση με την Ένωση και να στηρίξουν την ε, συνθήκη προσχώρησης. Είναι σημαντικό η Κροατία να λύσει τα διμερεί ζητήματα που έχει με κάποιες χώρες όπως η Σερβία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό των συνόρων, ε, τα αγνοούμενα άτομα και τους πρόσφυγες, καθώς και την επιστροφή περιουσιών. Ευχαριστούμε. Κύριε ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε ένα θέμα αρχής για την ένταξη της Κροατίας. Εγώ ψήφισα ναι, αλλά ψήφισα ναι μεν, αλλά η Κροατία ε, βεβαίω είναι ευρωπαϊκή χώρα, πράγμα που δεν μπορεί να πει κανεί για όλε τι υποψήφιε χώρε και βεβαίω θα πρέπει να έχει τη θέση τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμω, παραμένουν αρκετά προβλήματα στην Κροατία. Παράδειγμα, η διαφθορά μεταξύ άλλων. Και τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να λυθούν πρώτα, να αντιμετωπιστούν και να έρθουν σε αίσιο πέρας πριν ε, μπορέσει ουσιαστικά να ενταχθεί στην Ένωση ε, η Κροατία. Μόνο εφόσον πληρεί πλήρω τα ε, κριτήρια της Κοπεχάγης θα είναι σε θέση η Κροατία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη έκθεση του κυρίου Σουόβοντα για την αίτηση ένταξη Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Ανδρέας Σφάπ, πρώτος. Ε, κύριε Πρόεδρε. Οι ε, συνάδελφοί μου από τη Βάδη Βιτεμβέργη της Γερμανίας ε, ψηφίσαμε αποχή. Παρόλα αυτά ήταν πολύ μεγάλη η υποστήριξη και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου για το 28ο μέλος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Η ένταξη Κροατίας από την 1η Εβδόμη του 2012 δείχνει ότι παραμένει ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήταν πολύ αυστηρά τα κριτήρια που επιβάλαμε στην Κροατία και τα έχει καλύψει. Ωστόσο, πολλοί πολίτες ε, στην Ένωση θεωρούν ότι η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου θα πρέπει να είναι πολύ ε, αυστηρός και σοβαρός γνώμων και κριτήριο. Πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσει και τα κριτήρια. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να ενταχθεί η Κροατία θα πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές και ελπίζουμε την 1η Ιουλίου του 2012 να ενταχθεί πραγματικά ε, και ως πλήρες μέλος όταν θα έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Γι' αυτό με τους συναδέλφους ε, από το κρατήδιο της Βάδης Βερτεμβέργης αποφασίσαμε να ψηφίσουμε αποχή, αλλά με θετικό βλέμμα καλούμε την Κροατία να ξεπεράσει και τα τελευταία αναπομείνοντα εμπόδια. Ο κύριος Μικολάσικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κροατία εδώ και χρόνια προσπαθεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η πορεία οδήγησε σε μεγάλες αλλαγές στο δικαστικό σύστημα και στο αγώνα κατά της ε, διαφθοράς. Έχει επιτύχει πολλά η Κροατία, έχει επιτύχει μια πολύ καλή εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ε, σε πολλούς άλλους τομείς έχει κάνει τα απαραίτητα και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το πιο σημαντικό είναι φυσικά να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά στο επίπεδο του κράτους δικαίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό εγχείρημα και καθήκον για την Κροατία. Πρέπει εμείς να εργαστούμε, αποκοινούμε την Κροατία, ώστε οι κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματωθούν και από την Κροματία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι θα μπορέσει να γίνει η ένταξη της Κροατίας τον Ιούλιο του 2013. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ υποστηρίζω την πρόταση για την ιστοχή ε, της Κροατίας. Αλλά η Κροατία θα πρέπει να εργαστεί περισσότερο, θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να επιτύχει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να γίνει μέλος μονάχα όταν οι πολίτες της υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα και είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τις απαραίτητες προσπάθειες για μεταρρύθμιση. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, λειτουργία του δικαστικού τομέα και την αντιμετώπιση της ε, διαφθοράς. Επίσης, στον τομέα της αγοράς-εργασίας είναι απαραίτητο να γίνουν οι, οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, να περιοριστεί ο δημόσιος τομέας στην, στην Κροατία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε μια κατάσταση κρίσης. Θα πρέπει να προσαρμοστεί και η Κροατία και επίσης θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορέσει να βοηθήσει την ειρήνη στην περιοχή. Αυτό σημαίνει και για την ε, Σερβία και τη Μακεδονία πρέπει και αυτές να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ κύριο Χάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες όταν ανέφερε όταν ε, υπογράμμισε την ε, υποψηφιότητα για τις ε, εκλογές στην Κροατία, ο Σάσα Ράντοβιτς, ένας αγωνιστής υπέρ της διαφθοράς, συνελήφθη. Ήταν το κόμμα του το κόμμα της 21ης, του 21ου αιώνα και τόνισε ότι υπήρξε διαφθορά σε πάρα πολύ ψηλές θέσεις, σε πάρα πολύ υψηλούς κύκλους Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα επενδεδημένα συμφέροντα στο Ζάγκρεπ. Εγώ ήμουνα πρόσφατα στην, Κροατία και με λυπεί το πόσοι από τους γενναίους ανθρώπους της ε, Κροατίας είπαν ότι με τον τρόπο αυτό, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Ενώ στην πραγματικότητα οι διεφθαρμένοι θα βρουν ένα ευρώ ευρύτερο και λαμπρότερο πεδίο δόξας στη διαφθορά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κοινοβούλιο το οποίο εκλέγεται τώρα στην Κροατία είναι αυτό από το οποίο θα προέλθουν οι παρατηρητές στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως πρέπει να υπάρξει λοιπόν και κάποιος διεθνής έλεγχος τη στιγμή που φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο θα γίνει μια πολιτική λαθροχειρία. Ευχαριστώ κύριε Χάνεν. Περνάμε στην έκθεση Ραντ Κάι για την κοινοβουλευτική ασυλία του κυρίου Βίκτορ Ουσπάσκης το λόγο στον κύριο uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξέφρασα βαθιά διαφωνία με την ομάδα μου και καταψήφισα αντίθετα με την ομάδα μου σε ό,τι αφορά τα όσα συνέβησαν στο συνάδελφο Ουτσκάρσκι. Θα πρέπει να ακουστεί και άλλη πλευρά. Παραβιάστηκε αυτή η βασική αρχή. Η Λιθουανία είναι μια χώρα όπου συνεχίζονται υποτίθεται πολιτικές δίκες. Αυτό είναι άδικο ε, και παραπλάνηση. Είναι δημοκρατία η Λιθουάνια και βεβαίως υπάρχει το κράτος δικαίου για να εφαρμόζονται οι νόμοι. Δεν έχει σχέση με την περίπτωση Τιμοσέγκο στην Ουκρανία. Τι είναι αυτά τα παράλογα. Για ποιο λόγο να αποφύγει μια δίκη ένας πολιτικός που αφορά την τιμή του. Τι μήνυμα στέλνουμε στη χώρα μου για τη διάκριση των εξουσιών ότι είναι ανύπαρκτη στη Λιθουανία. Να τη, θα ήταν πραγματικά ε, σφάλμα να ε, έχουμε την ίδια αντιμετώπιση ε, στη Λιθουανία με την Ουκρανία και θα ήταν και λάθος για τη χώρα. Ευχαριστώ. Έκθεση Μπερές για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Και κατά πρώτο λόγο το λόγο έχει ο κύριος Δεάντζελης. Πρόεδρε, η κρίση δεν είναι πια μόνο απειλή, αλλά είναι ένα γεγονός που μπορεί να τροποποιήσει κοινωνικές και πολιτικές ε, καταστάσεις. Γι' αυτό και χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες. Η επιτυχία της στρατηγικής 2020 εξαρτάται από τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Τα κράτη-μέλη, ωστόσο, πρέπει να δουν την πολιτική, την οικονομική και τη δημοσιονομική τους ως κοινό ε, ε, συμφέρον και ενδιαφέρον. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε πιο μακριά. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο συντονισμό στην εφαρμογή εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων και στην αναχέτηση των φορολογικών απατών και της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο η στρατηγική 2020 να έχει μια περιφερειακή και κοινωνική διάσταση ε, μόνο μέσω της συμμετοχής των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους επιθυμητούς στόχους. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ελένα Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές ανισομέρειες με μια συμμετρική προσέγγιση, με μια πιο στενή συνεργασία. Όταν αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτή την ύφεση, αλλά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε θάρρος και υπευθυνότητα από την πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να εφαρμοστούν τα μέτρα λιτότητας που είναι απαραίτητα. Πρέπει να μειώσουμε λοιπόν τη διαφορά που υπάρχει σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρξει μια οικονομική ανάπτυξη. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει μια πρόβλεψη 1,5% σε οικονομική ανάπτυξη μέχρι το 2020. Δεν πρέπει οι προπολογισμοί μα να θέσουν ένα αμφιβόλο τη σταθερότητα όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και ο προπολογισμό των κρατών μερών να εναρμονιστεί. Όλα αυτά θα εξασφαλίσουν καλύτερη, καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. <laughs> κύριε Μπασέσκου και τώρα και πάλι ο κύριος Σιλβέστρος. Σας ευχαριστώ. Μία από τις επιπτώσεις είναι, της οικονομικής κρίσης είναι η αύξηση των ανισοτήτων ε, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει μακροοικονομικές ανισομέρειες ε, με συμμετρική προσέγγιση έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλεονάσματα τα υπερβολικά και τα ελλείμματα τα υπερβολικά. Συντονισμός οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και καλύτερη υποπτία των προπολογισμών. Τα σφάλματα που διαπράχθηκαν στα πρώτα δέκα χρόνια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματική Αποτελεσματικής Ένωσης έδειξαν ότι χρειάζεται πιο αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση που θα πρέπει να βασίζεται σε εποπτεία των κανόνων και πιο, πάγιο, πιο στέρεο μάλλον πρόγραμμα εποπτείας των εθνικών οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μέρφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μεσού σοβαρότερης κρίσης ε, της οικονομίας του καπιταλισμού στην Ευρώπη από το 30, η απάντηση των κυβερνήσεων είναι πολύ σαφής, μια λέξη λιτότητα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι η πλειονότητα των λαών στην Ευρώπη δεν συμφωνούν με τις λύσεις τους. Ο κόσμος γνωρίζει ότι πλούσιοι, όταν γίνονται πλουσιότεροι, η Ευρώπη ε, καταστρέφεται οικονομικά. Και γι' αυτό έχουμε το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Οικονομικής Εποπτείας είναι ένας τρόπος ε, αντιμετώπισης των ε, δημοκρατικών ελέγχων της δημοκρατικής νομιμότητας και ε, μέτρα που εφαρμόζονται στην Ιταλία και στην Ελλάδα με απικιακού τύπου τακτικές για λιτότητα. Βλέπουμε τι γίνεται στον ελληνικό προϋπολογισμό. Την άλλη εβδομάδα στην Τόλ, στη Βουλή μας, θα γίνει μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό μέχρι 4 δις γίνονται οικονομίες. Ε, είναι τεράστιες περικοπές αυτές και άγρια επίθεση στον Ιλλανδικό λαό. Και στο γερμανικό Bundestag ε, είδαμε τι αποφασίζεται. Αυτή είναι η οικονομική εποπτεία. Αυτό σημαίνει. Ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση. Για την ενιαία αγορά, ο κύριος ε, Λάιον έχει το λόγο. Κρίνει οπορτούνο Α, δεν θεώρησε μου να παραμείνει για να δώσει τις εξηγήσεις ο κ. Σιλβέστρης. Σε αυτή το πρώτο φόρουμ της ενίας αγοράς ε, κάλεσε την προσοχή όλων των επιπέδων, ε, των πολιτών, των ΜΚΟ, ε, και όλα αυτά για να ξεπεραστούν οι φραγμοί που συναντάνε περισσότερο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και επιβεβαιώνουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματική ευρωπαϊκή αγορά. 20 ε, χρόνια μετά τη δημιουργία της. Γι' αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε αυτή είναι το, το θέμα της αναγνώρισης των ε, επαγγελματικών προσόντων, την απόσπαση των εργαζομένων, καθώς και τα φορολογικά εμπόδια και τη λειτουργία ε, την ε, νομοθεσία όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες, ε, τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουν ούτως ή άλλως δοθεί πολλά πλεονεκτήματα στους πολίτες και σε 21 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρέπο έχει τώρα το λόγο για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε υπερψήφισα εγώ το ψήφισμα αυτό για το φόρμα της ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η ενιαία αγορά μπορεί ε, να είναι επωφελής με πολλούς τρόπους. Παρ' όλα αυτά, πολλοί πολίτες και πολλοί ε, επιχειρήσεις θα θεωρούν κάτι ξένο σε αυτούς τους καιρούς με κρίση χρέους, οικονομική και κρίση εμπιστοσύνης και έλλειψη θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να πεισούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής ενέας αγοράς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε τρόπο στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουμε τα μέτρα που συμφωνήθηκαν. Η εσωτερική αγορά παραμένει από τα σημαντικότερα και καλύτερα επιτεύγματα της Ένωσης και ε, παράγουν σταθερότητα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Τελευταίο θέμα. Με επεξηγής ψήφου έχει να κάνει με την πρόταση ψηφίσματος για την παγκόσμια απάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για το AIDS. Και πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Σιμάνσκι. Ε, Panie Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ένταση όλων των δράσεων για την καταπολέμηση του HIV και του AIDS είναι πολύ σημαντική και σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο ένωσης. Οι ε, προτάσεις που ακούσαμε και τα ψηφίσματα για το AIDS ε, βεβαίως αξίζουν οπωσδήποτε την υποστήριξή μας, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας. Δυστυχώς, ο συνήθως, όταν ε, πρόκειται για ζητήματα υγείας, οι προτάσεις που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνουν και την προαγωγή των αμβλώσεων. Γι' αυτό εγώ το καταψήφισα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την εξαίρετη έκθεση ε, και το Εργατικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, σφαιρική και ε, η ε, σεξουαλική ζωή της γυναίκας και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχει πρόσβαση κάθε γυναίκα στην αντισύλληψη και της εκτάκτου ανάγκης και όπου χρειαστεί αμβλώσεις, ναι. Θα πρέπει να ε, ε, δοθεί έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα και την καλωσορίζουμε. Επίση, χαιρετίζουμε τις τεράστιες θετικέ εξέλιξεις. Όπως είπα και στην αρχή της συζήτηση, θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απελευθερώσει, να ξεπαγώσει τα κονδύλια για το Παγκόσμιο Ταμείο ε, του AIDS. Σε αντίθεση με το προηγούμενο Βρετανό ομιλητή, πρέπει να πω ότι η υποστήριξη των ε, οικουμενικών ε, δικαιωμάτων ε, δεν είναι ε, απεικιοκρατικό, είναι ουσιαστικό για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους. Ο κύριος Σιλβέστρης. Θετικά δέχομαι, Πρόεδρε, το κείμενο αυτής της πρότασης ψηφίσματος που εκφράζεται θετικά για έναν από τους στόχους της χιλιετίας όπως προκύπτει από τις στατιστικές ε, μιας παραγράφου της έκθεσης που υπερψηφίσαμε, η μόλις αφορά περισσότερο νέους και γυναίκες αυτή τη στιγμή. Η εκστρατεία για την ενημέρωση για το ιό του HIV ήταν πολύ έντονη το 80, τη δεκαετία του 80, ενδιαφέρον για αυτή την ε, ασθένεια σιγά σιγά έχει εξασθενήσει. Λες και ο κίνδυνος δεν υπάρχει πια. Θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ε, πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος που, έχει, που είναι οροθετικός δεν έχει απαραίτητα το AIDS ή ότι δεν υπάρχει ε, τεστ για το AIDS αλλά για το νιό HIV. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενημερωθεί ένα θέμα το οποίο, στο οποίο πολλά μπορούμε να πούμε και να ενημερώσουμε προσπαθώντας να βρούμε γενική απάντηση στο θέμα μέσω της καλύτερης γνώσης και ενημέρωσης του κόσμου. Ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστρη. Στο λόγο έχει ο κύριος Μέρφη. 33 εκατομμύρια άτομα ζουν σήμερα με τον ιό του AIDS και 3 εκατομμύρια ε, μολύνονται κάθε χρόνο, 2 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο. Φαίνεται ότι θα γίνει στον 21ο αιώνα ο κύριος αίτιος θανάτου. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική απάντηση σε αυτή την αρρώστια. Δυστυχώ από πολλέ απόψει πηγαίνουν προ τη λανθασμένη κατεύθυνση. Τα προγράμματα καταπολέμησης του AIDS έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση κατά 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μεγάλες περικοπές που γίνονται σε δημόσιες υπηρεσίες έχουν εισαχθεί ε, και μέτρα Λιτότος για τα φάρμακα κατά του AIDS που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων. Έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι σε ό,τι αφορά την καλύτερη πρόσβαση και τα καλύτερα φάρμακα κατά του AIDS, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν. Η ύπαρξη ευαισθητεχνιών που προστατεύουν τη φαρμακευτική βιομηχανία εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Πρέπει να εθνικοποιηθούν λοιπόν οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και να υπάρξει μια σημαντική υποστήριξη σε παγκόσμια έρευνα χωρίς ευρεσιτεχνίες για να βελτιωθούν τα φάρμακα για όλους. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο κύριος Φιλιπ Κλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση για το HIV και το AIDS. Όχι γιατί έχω πρόβλημα ε, να έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και περίθαλψη οι οροθετικοί και οι άρρωστοι με το AIDS, ούτε για τα φάρμακα. Αυτό το πρόβλημα που έχω είναι ότι έχουν παρισφρήσει πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό θέμα. Παράδειγμα, παράγραφος 22, όπου ζητούν και παραθέτω ε, ασφαλή και νόμιμη άμβλωση τέλος της παράθεσης. Τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακατεύεται σε τέτοια θέματα. Αυτό είναι ζήτημα των κρατών μελών. Και αν υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν νόμιμες αυλώσεις, θα πρέπει να είναι σε θέση να το πραγματοποιούν. Επίσης, ζητούν για τα δικαιώματα, ε, την ιδιωτική ζωή ε, των αρρώστων. Εντάξει είναι αυτό, αλλά δεν γίνεται λόγος για το πώς εκείνοι που έχουν επαφή με ασθενεί από AIDS ε, προστατεύονται. Γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλεύτριε, όταν δεν ξέρουν ότι ε, είναι ασθενεί ή οροθετικοί ασθενεί τους. Και η κοινωνία θα ε, πρέπει να μπορεί να προστατεύεται, όχι μόνο οι άρρωστοι. Ευχαριστώ κύριε Κλάης. Με την παρέμβαση αυτή ολοκληρώνεται ο γύρος των επεξηγήσεων ψήφου. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν το λόγο. και που τηρήσατε και τους χρόνους. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε ουσιαστικά να διακόψω κανέναν ε, παρεμβαίνοντα. Έχω λάβει από το Συμβούλιο δύο κοινέ θέσει για πρώτη ανάγνωση, ε, καθώς και τους ε, λόγου που του οδήγησαν να το εγκρίνουν μαζί με τι αντίστοιχε θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τίτλοι θα ανακοινωθούν στα πρακτικά τη παρούση συνόδου και η τρίμηνη προθεσμία που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφανθεί αρχίζει από αύριο 2 12